θα υποβληθούν ή στην, ε, για, για έγκριση στο Κοινοβούλιο την επόμενη ε, ολομέλεια και όλα τα ε, ψηφίσματα θα αποσταλούν στους αποδέκτες του.